Και να σας ανακοινώσω κύριε και κύριοι ότι ε, έλαβα και ένα αίτημα γραπτό για την κατάργηση των γραπτών αιτημάτων. Αλλά είναι μη παραδεκτό αυτό σύμφωνα με τον κανονισμό. Οι επιτροπές λοιπόν δημοσίευσαν πέντε κείμενα του Κοινοβουλίου και εάν έως 24, εως 24 ώρων δεν λάβω οποιαδήποτε ένσταση από κάποια πολιτική ομάδα θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Τους τίτλους λοιπόν των ε, ψηφισμάτων των ε, νομοθετημάτων αυτών θα τους βρείτε στα πρακτικά της κυβέρνησης. Ε, σύμφωνα με την κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία, λοιπόν,